Bene, colleghi, diamo inizio subito, abbiamo molti punti. Έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 9, το σημείο 9 της ημερήσια διάταξης, ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό 73-2009 ε, όσον αφορά το ημερολογικό έτος 2003. η ε, Εισηγητής Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε για την πρόταση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μείωση κατά 5% των άμεσων ενισχύσεων για τις φετινές αιτήσει των γεωργών, χαμηλώνοντας στο μέγιστο τον πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, το οποίο το που τα διαπραγματεύτηκαν ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις 7 και 8 του περασμένου Φεβρουαρίου. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε καμιά συνεννόηση με το Συμβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 16 ε, τροπολογίες στην Επιτροπή Άγκρη. Πρέπει να εξετάσουμε και να ψηφίσουμε τις πέντε τροπολογίες που υπέβαλε η Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό στη γνωμοδότησή της. Δεν ξέρω, ο Λουίς θέλει να πάρει το λόγο πρώτα. Όχι. Αν είστε όλοι έτοιμοι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αμέσως με την ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε με την τροπολογία. Μπορούμε διανατάσσεως της χειρός. Τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Συνάδελφοι, υπάρχει διχογνωμία. Νομίζω θα πάμε ηλεκτρονικά. Ε, ζητώ συγγνώμη. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 2 του εισηγητή. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Okay. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 13, Νταντέν. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Είμαστε όλοι υπέρ. Εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να μην κάνουμε λάθος, συνάδελφοι. Υπέρ οι περισσότεροι. Εντάξει, με πλειοψηφία, άνετη. Ε, ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 16, Lion Πόλσεν. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επί της 16, Lion Πόλσεν. Ψήφισαν όλοι. Ευχαριστώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με πλειοψηφία. Στη συνέχεια θα ψηφίσουμε τη 14 14. Αντρόβε και άλλοι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Και θα έλεγα... Α, απορρίπτεται. Ισοψηφία. Και τώρα θα ψηφίσουμε... Την τροπολογία 1 του εισηγητή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Αρχίζει, έχει αρχίσει. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Και έχει εγκριθεί με πολύ άνετη πλειοψηφία. Στη συνέχεια, οι δύο τελικές ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία. ελπίζω υπέρα, πέρα της ψηφοφορίας και τελική ψηφοφορία το νομοθετικό ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας. Συνάδελφοι, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο και την Προεδρία θα αναλάβει ο Αντιπρόεδρος Σεκελέσκη. Πρέπει να φύγω γιατί έχω μια συνάντηση. Θέλω να πω ότι μετά από τη συζήτηση που είχαμε χθες με τον Επίτροπο Τσόλος, για το επίμαχο θέμα του παρθένου ελαιόλαδου, του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, θα το θυμάστε, και μετά από αίτηση πολλών ε, συναδέλφων της Επιτροπής έγραψα μια επιστολή και ζήτησα εξ ονόματος της Επιτροπής μια επίσημη απάντηση από τον Επίτροπο πάνω στο θέμα της υποχρέωσης χρήσης μη ανακυκλώσιμων φιαλών για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα εστιατόρια. Ε, και ζητώ από τον Επίτροπο να λάβει απόφαση επί του θέματος αυτού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ε, γιατί δεν θέλουμε να μένει αυτή η εμφιβολία πάνω σε, σε μια διάταξη για την οποία υπήρξαν πολλές διχογνωμίες και μεγάλη συζήτηση. Οπότε, αν δεν υπάρξει κάποια αντίθετη εξέλιξη, γράφουμε αυτή την επιστολή προς τον Επίτροπο και λέμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε διαβάσει μόνο πληροφορίες στα άρθρα των εφημερίδων. Ε, δεν ε, συμμετείχαμε στη διαδικασία. Λοιπόν, συνάδελφοι, αφήνω την Προεδρία εδώ στον Αντιπρόεδρο και σας αφήνω. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο ο Πρόεδρος. πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση. Ο Ζωζέ Μποβέ είναι ο εισηγητής ε, για τη γνωμοδότηση, ο συντάκτης. Υπάρχουν 62 ε, τροπολογίες πάνω σε αυτή την γνωμοδότηση για την επικύρωση του πρωτοκόλου Ναγκόγια. 35 κατατέθηκαν από τον ίδιο τον κύριο Ζωζέ Μποβέ, τον οποίο και δίνω τον ε, λόγο. Ε, δεν θέλει να λάβει το λόγο ο, Ζωζέ Μποβέ, οπότε ας περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Καταρχήν. Poprawka 10. Otwieram Λοιπόν, τροπολογία υπαριθμών 10, ε, ψηφίζουμε. Zamykam głosowanie. 33 do 30, 21. Έκλεισε η ψηφοφορία. 31 υπέρ. Άρα δηλαδή εγκρίνεται. Πάμε στο 47. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πάμε στο 11. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 48 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. 12 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 17 κατά. Απορρίπτεται. Επόμενη ψηφοφορία για το 49. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 21 ψήφους υπέρ. Πρόεδρε, Κοιτάξτε, υπήρχε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη μετάφραση γιατί Μα είπαν ότι ψηφίζαμε για την 13 ενώ ψηφίζαμε για τη 49. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Και το πρόβλημα είναι ότι η μετάφραση από τα πολωνικά ε, αργεί λιγάκι. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να προχωράτε λίγο πιο αργά. Głosowanie 13. 13. Kto Εντάξει λοιπόν για το 13. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Τροπολογία 13. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. «26 υπέρ». Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τη 49 και τη 14. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 παρακαλώ ψηφίζουμε για τη 15 παράγραφο, ε, τροπολογία 15 έκλεισε η ψηφοφορία Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 16. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με 21 ψήφους κατά. 17 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 18. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 19. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ο κ. Κάπουλας. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά διαπιστώνω ότι αυτό που ε, φαίνεται στην οθόνη είναι η επόμενη τροπολογία από αυτή που ψηφίζουμε. Δεν ξέρω τελικά το σύστημα λειτουργεί ή όχι. Όταν είπατε, παραδείγματο χάρη κύριε Πρόεδρε, ότι ψηφίζουμε την τροπολογία 16, εμφανίστηκε 17 στην οθόνη. Το σύστημα δεν λειτουργεί. Τι γίνεται. Κάθε φορά που ψηφίζουμε αυτό είδα. Να βγαίνει η επόμενη τροπολογία, όχι αυτή που ψηφίζουμε. Κύριο Σταραμπελά, νομίζω ότι είναι διαφορετικό το σύστημα στην Επιτροπή από ότι στην Ολομέλεια που ανακοινώνεται παράγραφος και τροπολογία. Εδώ μπαίνουν τροπολογίες με τη σειρά. Ε, που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορίας. Άρα το νούμερο ε, που βλέπουμε στην ε, οθόνη δεν έχει να κάνει με την τροπολογία, δεν είναι ο αριθμός της τροπολογίας και πρέπει να προσέχετε την εκφώνηση από τον πρόεδρο κάθε φορά. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε για την 20 παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 20. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Για την 50. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 51. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 52. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22. Ψηφίζουμε για την 22 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Για την 23 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 53. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 55. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Για την 24, ψηφίζουμε για την 24, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25 ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται 18-15 το αποτέλεσμα 56 ψηφίζουμε για την 56 έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 26. Για την 26 παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 26. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία, έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται. Για την 27. Προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία μετά τις συζητήσει που είχαμε για τις προθεσμίες σε σχέση με το αρχικό κείμενο που έλεγε ότι διαβιβάζουν οι αρμόδιες αρχές στην Κομισιόν τις πληροφορίες που έχουν λάβει κάθε δύο χρόνια κτλ. κτλ. Εμείς προτείνουμε για να είμαστε σύμφωνοι με τις περισσότερες πολιτικές ομάδες και για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια να αναδιατυπωθεί το κείμενο και να λέει ότι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν τις πληροφορίες ε, που έχουν δοθεί και τις διαβιβάζουν τους προθεσμίες έξι μηνών. Αυτό ε, συνάδει ε, με ό,τι έχουμε και μετά λέμε ότι τις πληροφορίες που έχει λάβει η Κομισιόν μέσα σε έξι μήνες τι διαβιβάζει για την έγκριση του πιστοποιητικού μας κτλ. Δηλαδή, αντί για δύο χρόνια, ουσιαστικά θέλουμε να περιορίσουμε, να συντομεύσουμε την προθεσμία και να την κάνουμε έξι μήνες. Συμφωνείτε με αυτή την προφορική τροπολογία. Ωραία, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 27 με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 27, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28, κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα. 20 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Είκοσι υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Το εισηγητή υπέρ. Α, μάλλον άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται. Τροπολογία 57 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασο. 27 προς 6. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασο. Εγκρίνεται το προς 14. τροπολέγια 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ και καμία ψήφος κατά. Επόμενη, 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται 7 προς 25 τροπολογία 59 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 16 προς 9 τροπολογία 32 άρχεται η ψηφοφορία Εγκρίνεται. 26 6 κατά. Τροπολογία 32. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Όχι, λάθος. Τροπολογία 60. Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 60. Έλξη ψηφοφορία εγκρίνεται 18 προς 11. Το πρωί 61 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 16 προς 14. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται 31 υπέρ 1 κατά η ψήφη 34 άρχεται ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται 15 προς 16 62 άρχεται ψηφοφορία πέρασε Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 27 υπέρ, 5 κατά εγκρίνεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 23 προς 7 εγκρίνεται 36 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 21 7. 37 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα 23 προς 7 εγκρίνεται τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι, λάθος. Δεν ψηφίζουμε τη 2. Πάμε στην 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 15 προς 16, 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 29 προς 2. Τροπολογία 39. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 προς 45. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. 44, συγγνώμη. 44. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται, επαναλαμβάνω. Τροπολογία 45, έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 25 προς 6. Τροπολογία 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 25 προς 6. Και τώρα ψηφίζουμε την ομοδότηση με τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Και ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Ζωζέ Μποβέ. Περνάμε στο σημείο 11, που είναι το πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκη και ισότιμη συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους το οποίο πρωτόκλοπη συνάπτεται στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. δεν έχουν τροπολογίες, ε, προτείνει να εγκρίνουμε ε, το πρωτόκολλο κύριος ε, Μποβέ. Μπορούμε να σφισουμε δηλαδή υπέρ ή κατά. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Α, όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια και τώρα περνάμε στο σημείο 12, το επόμενο σημείο της διάταξης. Προϋπολογισμός 2014 εντολή για τον τριμέρι διάλογο. Κανονικά θα έπρεπε τώρα να ε, συζητούμε τον προπολογισμό, αλλά στα τέλη Μαΐου και όχι στα τέλη Απριλίου παρουσιάζει η Κομισιόν φέτος τον προπολογισμό της. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, εκπονήσουμε την γνωμοδότησή μας για την εντολή για τον τριμμένο διάλογο όπως ε, κάναμε συνήθως, απλά κατευθείαν τις τροπολογίες για την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών. Για την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, σε ό,τι αφορά πιλωτικά προγράμματα και προπρασκευαστικές δράσεις, 4 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την Βασιλίτσα Βιόριτσα Ντάντσιλα. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați specificat, Comisia Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είχε προτείνει μέχρι τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όπω είπατε, το σχέδιο προπολογισμού για το 2014. Αποφάσισε όμω να αναβάλει την υποβολή της πρότασης αυτής. Άρα ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ε, ένα έγγραφο από την Κομισιόν και είναι ε, επίγουσα και ασαφής η κατάσταση. Ο πρόεδρος, μάλλον ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι θα κάνει την πρότασή του στην Επιτροπή Πρόεδρων σήμερα, όμως ο μας, του 2014 ε, ακόμα τε, τε, τελεί υπό αναβολή. ό,τι αφορά τις συζητήσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σας ενημερώνω ότι ο Επιτρόπος Λεβαντόφσκι χρησιμοποιεί τα ποσά που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, αλλά τα ποσά αυτά, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα απέρριψε το Κοινοβούλιο. Επομένως, η Επιτροπή Άγκρη δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θα καταθέσουμε μόνο τροπολογίες απευθείας ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όταν θα έχουμε ποσά για το 2014. Νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει να προετοιμάσει το προπολογισμό του 2014 πάνω σε ρεαλιστικές βάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2014-2020, χωρίς να βασιστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8η και 9 ης γιατί όπως είπα, έχει ε, απορριφθεί από το Κοινοβούλιο η πρόταση του Συμβουλίου. Αν είναι ανεπαρκής ο προπολογισμό, ε, θα περιπλακεί η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Δεν θα μπορεί να είναι ρεαλιστική. Και όπως είδαμε χθε, απομένουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν μπόρεσαν να, να λυθούν. Εδώ πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2014 είναι μεταβατική χρονιά. Είμαστε μεταξύ δύο πολιτών δημοσιονομικών πλαισίων. Είναι και ε, χρονιά μετάβασης και για την Ευρωπαϊκή Γεωργία προς μια πιο δίκαιη οικολογική γεωργία που θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές καταστάσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν μειωθεί ο προπολογισμό του 2014, το αποτέλεσμα θα είναι να επιδεινωθούν οι ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των Ευρωπαίων αγροτών και μεταξύ των διαφόρων αγροτικών περιοχών. Εμείς αντιλαμβανόμαστε και τι οικονομικές και τις δημοσιονομικές δυσκολίες αυτό, όμω δεν σημαίνει κατά ανάγκη μείωση του προπολογισμού για τη γεωργία. Πιστεύω ότι το 2014 θα πρέπει να είναι η χρονιά κατά την οποία οι αγρότες θα δουν την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ όχι ως φορτίο βάρος, αλλά ως ένα πραγματικό εργαλείο ενίσχυσης των συστημάτων που θα τους δώσει σωστές, καλές απαντήσεις. Ο γεωργικός προπολογισμό και ο προπολογισμό ανάπτυξης της υπαίθρου για το 2014, παραλαμβάνω, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης και μεγαλύτερου θετικού αντικτύπου της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει να εξασφαλίζει και ένα κανοποιητικό ε, βιωτικό επίπεδο για τους αγρότες για τις πιλωτικές, ε, πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουμε την προθεσμία της 4ης Ιουνίου, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε. Και αφού δεν έχουμε ακόμη περιπολέξουμε για το 2014, ενδέχεται να αλλάξει αυτή η προθεσμία. Αφού η Κομισιόν ήδη ανέβαλε την παρουσίαση του προπολογισμού. Υπάρχει ένα έγγραφο ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπασκευαστικέ δράσει. το οποίο ε, επισυνάπτεται στο σχέδιο του προπολογισμού συνήθως, φέτος δεν το λάβαμε ακόμα. Όλα τα έντυπα που έχουμε λάβει για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να τα λάβουμε και να τα μελετήσουμε. πρέπει να έχουμε ενημέρωση και πρέπει και στο μέλλον να υπάρχει καλύτερη θεσμική ε, διοργανική συνεργασία για να μπορούμε πιο επικοδομητικά να συνεργαζόμαστε, να έχουμε καλύτερες, πιο αναλυτικές πληροφορίες στη διάθεσή μας που θα τις λαμβάνουμε έγκαιρα από την Κομισιόν. Νομίζω οι συνάδελφοι συμμερίζονται τις απόψεις μου γιατί τα συζητήσαμε χθε και με τον αρμόδιο τη Γεωργία Επίτροπο. Στόχος μας είναι μεγαλύτερη ε, διαφάνεια, ορατότητα και πιο σαφείς, ξεκάθαρες αποφάσεις από την Κομισιόν και από την Επιτροπή Άγκρη. Ευχαριστώ και περιμένω τις συστάσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση. Παρακαλώ πολύ. Rozumiem, Οι εξηγήσει που δώσατε ήταν τόσο εκτενείς και αποκαλυπτικές που από ό,τι φαίνεται ε, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Αλλά ας δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος μας μοιάζει να μην είναι εδώ παρόν. Ε, είναι άλλη, μια άλλη κυρία όμως εδώ από την Επιτροπή. The... Ε, δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Το σχέδιο του προϋπολογισμού κάποια στιγμή θα ε, δημοσιευτεί. Νομίζω αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα εξετάσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πιλωτικά προγράμματα που θα καταθέσετε ως Επιτροπή. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνω το λόγο και στην εισηγήτρια. Ε, ο σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Βοητσοκόφσκι, είναι εδώ. Προτείνω μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις εργασίες μας πιο αποτελεσματικά. Να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 2014 μέσω τροπολογιών που θα υπολοιθούν απευθείας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Możemy Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόταση. Οι τροπολογίες πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 4 του μηνός, αν κατάλαβα καλά. Όχι, όχι, έλεγα ότι δεν έχουμε το σχέδιο για το 2014 και πρότεινα την επόμενη εβδομάδα να κανονίσουμε μια συνάντηση με το σκιώδη εισηγητή για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από κοινού για την υποβολή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Επιτροπή προπολογισμού όταν με το καλό μας έρθουν τα έγγραφα. Ε, Εντάξει, πολύ ωραία προφανώς και συμφωνούμε με αυτό που μόλις τώρα είπατε. Πάμε τώρα στα σημεία 14 έως 17 ε, που θα τα εξετάσουμε από κοινού όλα μαζί. Είναι τα μέτρα, ε, προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Η Επιτροπή στις 6 Μαΐου ενέκρινε ένα πακέτο ε, για να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα όσον αφορά στην προστασία της υγείας. Μιλάμε για περίπου 70 νομικές πράξεις και αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο ε, θέλει να περιορίσει τον αριθμό των διατάξεων σε ε, τέσσερις. Η δική μας λοιπόν επιτροπή είναι η καθήλυνα αρμόδια για τα εξής θέματα μέτρα κατά των ε, επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά, κυρίως ε, όσον αφορά στο πολλαπλασιαστικό υλικό και στην προστασία των ζώων, την ε, γνωμοδότησή μα, ε, θα την εκπονήσουμε για τα εξή θέματα. Έλεγχη και δραστηριότητε που πρέπει να λάβουν χώρα έτσι ώστε να εφαρμοστεί το δίκαιο για τα τρόφιμα ε, και τις ζωοτροφές. Κατόπιν ε, είμαστε αρμόδιοι για το πολυπλασιαστικό υλικό, για την υγεία των φυτών και για τα προστατευτικά υλικά, ε, προστατευτικό υλικό των ζώων. Εγώ προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, παρουσιάσει και τις τέσσερις αυτές προτάσεις και μετά θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Ο κύριος Φαν παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Φαν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το πακέτο για, τις, για τα πιο ασφαλή τρόφιμα στην Επιτροπή σας σήμερα. Με την άδειά σας θα κάνω πρώτα μια γενική επισκόπηση και στη συνέχεια θα ζητήσω από τους συναδέλφους να παρουσιάσουν τις ειδικότερες λεπτομέρειες της κάθε πρότασης. Το πακέτο αυτό των τεσσάρων προτάσεων είναι η συνεισφορά μας για την ενοποίηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το σύνολο της τροφικής αλυσίδας. Δεν προτείνουμε να επαναεπινοήσουμε τον τροχό. Θέλουμε απλώς να απλοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε την νομοθεσία μας με σαφή έμφαση στην πρόληψη και μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία ελπίζουμε θα επιφέρει άμεσα ωφέλη στον σχετικό τομέα, στους καταναλωτές και στη διοίκηση, στις διοικήσεις των κρατών μελών που πρέπει να υλοποιήσουν τους κανόνες αυτούς. Είναι ξεκάθαρο ότι η γεωργική παραγωγή και η αλυσίδα της τροφής συνολικά έχουν κέρια σημασία για την κοινωνία σε αυτούς τους καιρούς της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δυστοκίας. Ε, ο ρόλος της νομοθεσίας είναι να παρέχει κατάλληλα εχέγγυα, όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και προς το συμφέρον των τομέων, των παραγωγικών τομέων. Η τομεί αυτή, ο γεωργικός τομέας, όπως γνωρίζουμε από προηγούμενη εμπειρία, τόσο στην φυτοπαραγωγή όσο και στη ζωοπαραγωγή και στην παραγωγή και διανομή, κατανομή των τροφίμων, πλήγεται έντονα από την απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και από τις επιπτώσεις της ε, κρίσης. Παρόλο που η κρίση δεν έχει πάντοτε κάποιο περιεχόμενο ανασφάλειας ή κινδύνου των τροφίμων, ε, πρέπει να προστατέψουμε την ακαιρεότητα του συστήματος, γιατί υπάρχουν και επιπτώσεις διεθνούς εμβέλειας. Οι πιο απλοί κανόνες θα μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε και να υπεραμεινθούμε του συστήματό μας στις συζητήσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους. Οι σωστοί μηχανισμοί αντίδρασης σε έκτακτες περιπτώσεις θα επιτρέψουν στο σύστημα να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των εταίρων μας στο δικό μας σύστημα. Η σύγκληση των κανόνων με τα διεθνή πρότυπα ε, θέτει, μια, θέτει στέρεα θεμέλια για τις εμπορικές μας σχέσεις η συμβολή μας στην περαιτέρω εξέλιξη αυτών των κανόνων ε, γίνεται ευνοϊκά αποδεκτή ε, στο διεθνές περιβάλλον. Ο σκοπός μας είναι να εξοπλιστούμε με τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις που μόλις περιέγραψα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεών μας για την υγεία των ζώων και των φυτών είναι η έμφαση στην πρόληψη οι, ουσιασ... διατάξεις ουσιαστικού δικαίου θα συμπληρωθούν από μια χρηματοδοτική πρόταση η οποία βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και θα καθορίσει την ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δοθεί προς τα κράτη-μέλη για να εξαλείψουν κινδύνους κατά της ε, υγείας και της ζωής ζώων και φυτών. Συγκεκριμένα, για την ε, υγεία των ζώων, Στόχος μας είναι μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του εμβολιασμού ως εργαλείου και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη μετακίνηση και τη μεταφορά των ζώων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για την υγεία των φυτών έχουμε ένα νέο σύστημα εποπτείας το οποίο θα βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε νωρίτερα τους επιβλαπείς οργανισμούς και να αντιδρούμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Είναι σαφές ότι πρέπει να εστιαστούμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας εκείνους τους επιβλαβείς οργανισμούς που έχουν σημασία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θέσουμε τα κατάλληλα μέσα στη διάθεση των κρατών μελών για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς το κοινό συμφέρον. Η μείωση και πάλι του διοικητικού φόρτου είναι ένας στόχος μας στην απλοποίηση ε, του συστήματος μεταφοράς ε, των φυτών έτσι ώστε να διευκολύνεται η χνηλασιμότητα. Όπως ξέρετε η χνηλασιμότητα αποτελεί βασική αρχή πλέον του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων. Για το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών ε, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, τις οποίες ίσως και εσείς αντιληφθήκατε πρόσφατα. Υπάρχει μια ανησυχία ότι η Επιτροπή ε, προτιμά τους παραδοσιακούς ε, πολλαπλασιαστές και ιδίως για την οργανική γεωργία και ο διοικητικός φόρτος ε, θα είναι σε βάρος των μικρών παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού και σε βάρος των πιο σπάνιων ειδών. Αναγνωρίζουμε την, ε, τις μικροεπιχειρήσεις ε, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θύλακες της αγοράς, ε, οι οποίες απολαμβάνουν μεγάλων εξαιρέσεων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι διάφορες τάσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για βιώσιμη γεωργία, η διαφύλαξη των φυτικών γενετικών πόρων θα αναγνωρίσουν και το σύστημα των ποικιλιών, της καταγραφής ποικιλιών, της καταχώρησης ποικιλιών και ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανοιχτή πρόσβαση σε ποιοτικά και υγιή υλικά στους επίσημους ελέγχους υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων. Η ε, έλεγχη στα σύνορα, ε, οι εξαιρέσεις προς τις μικροεπιχειρήσεις ε, είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Σημασία έχει επίσης να αντλήσουμε τα διδάγματα από, τα πρόσφατα, από τις πρόσφατες εξελίξεις τις κυρώσεις από την εισαγωγή υποχρεωτικών προγραμμάτων ελέγχων, όπως ξέρετε για το, για το αλογίσιο κρέας. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η πρόταση που έχετε μπροστά σας και το κείμενο και οι χρηματοδοτικές πτυχές που θα έρθουν σε γνώση σας σύντομα ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Σίγουρα θα θέλετε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο γύρω από τις αρχές που σας προτείνουμε και αργότερα γύρω από τις λεπτομέρειες των εφαρμοστικών πράξεων. Ε, συμμερίζομαι όλες σας τις ανησυχίες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θέλουμε οι μελλοντικές τεχνικές λεπτομέρειες να προκύπτουν μετά από κριτική εξέταση των κανόνων που έχουμε στα χέρια μας. Όπως είπα, δεν θέλουμε να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Ε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλογο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να σας προ... παρέχοντάς σας διασαφηνίσεις, επεξηγήσεις και βοηθώντας σας στη συζήτησή σας. Η Ιρλανδική και η Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου επενδύει έντονα στα θέματα αυτά. Από την πλευρά μας ελπίζω ότι το κείμενο που έχετε στη διάθεσή σας θα σας βοηθήσει ε, στο μέλλον, στο νομοθετικό σας έργο και στις ε, ανταλλαγές απόψεων με τα άλλα όργανα. Και τώρα, με την συμφωνία σας, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω από τους συναδέλφους να παρουσιάσουν τις τέσσερις προτάσεις κατά τη σειρά που γράφονται. Πρώτον, επιβλαβείς οργανισμοί. Δεύτερον, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών. Τρίτον, υγεία των ζώων. Και τέλος, η έλεγχη. Δίνω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για το κάθε ντοσχέ. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ε, παρακαλώ, επόμενος ε, συναδελφός σας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν τον ε, κανονισμό ε, για τα προστατευτικά μέτρα που θα προστατεύσουν την υγεία των φυτών. Όπως αναφέρθηκε στην ε, προηγούμενη παρέμβαση, ο δικός μας ο κανονισμός ασχολείται κυρίως με την πρόληψη την προστασία των εσοδιών της γεωργίας, της δασοπονίας ε, την προστασία τους από επιβλαβείς οργανισμούς που θα μπορούσαν να διεισδύσουν στην επικράτειά μας. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί σε άλλες ε, πύρους, ε, που είναι πολύ επικίνδυνοι. Εδώ δεν υπάρχει αντίσταση στην Ευρωπαϊκή πύρο και όλοι αυτοί οι οργανισμοί θα μπορούσαν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Εσοδιά. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα καλό καθεστώς ε, για την προστασία των ζώων. Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που βασίζεται στην οδηγία του Συμβουλίου 2000 ε, αυτό το καθεστώς ε, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης και αυτοί οι οργανισμοί πλέον μπορούν να διεισδύσουν στην Ευρώπη και να καταστήσουν τα οικοσυστήματα και τις εσοδιές περισσότερο τροτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να υπάρξει μια νέα άποψη και αυτή την έχουμε διαμορφώσει, σας την έχουμε καταθέσει Και γι' αυτό εμείς ε, αποφασίσαμε να ρυθμίσουμε τα θέματα των επιβλαβών οργανισμών ε, που θέλουμε να κρατήσουμε μακριά από την Ευρωπαϊκή Επικράτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του κανονισμού. Θα εστιάσω την προσοχή μου σε τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η πρόληψη. Πρόληψη απέναντι σε νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτή λοιπόν η προληπτική προσέγγιση εφαρμόζεται σε δύο επίπεδα. Στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σημεία εισόδου σε αυτήν. Ας δούμε το πρώτο. Εκεί γίνεται κατηγοριοποίηση των επιβλαβών οργανισμών, των φυτών και κάθε κατηγορία συνδέεται με εναρμονισμένα μέτρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτά οι οργανισμοί που πρέπει να μπουν σε καραντίνα και πρέπει να κρατηθούν ε, μακριά από την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τα, οι υπόλοιποι επιβλαβείς οργανισμοί που ήδη έχουν εμφανιστεί εδώ αλλά επηρεάζουν τους σπόρους, τα φυτά προς ε, φύτευση. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε διάφορες ε, κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο που συνεπάγονται. Έχουμε ε, επιβλαβείς οργανισμούς ε, πρώτης προτεραιότητας, αυτοί που πρέπει να μπουν σε καραντίνα, που έχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Και ε, λόγω ακριβώς αυτών των προεκτάσεων εκεί πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες, να κατατίθενται ετήσιες ε, μελέτες, ε, να υπάρχει ετοιμότητα δράσης από πλευράς κρατών μελών να υποβάλλονται εκθέσεις από τα κράτη-μέλη για κάθε μία κατηγορία αυτών των επιβλαβών οργανισμών και όλα αυτά να συνδέονται και με ενισχυμένη συγχραματοδότηση δηλαδή την αποζημίωση των ε, εμπόρων ε, στην περίπτωση που πλήττεται η εσοδιά τους από αυτούς τους οργανισμούς. Ένα άλλο μέτρο που προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιβάλλουμε μια προληπτική προσέγγιση. Ένα άλλο μέτρο είναι τα προγράμματα πολιτών ε, ερευνών και η συγκέντρωση πληροφοριών. Τα κράτη-μέλη μπορούν να διεξάγουν τέτοιου είδους έρευνες για να διαπιστώσουν κατά πόσον υπάρχουν τέτοιου είδους επιβλαβείς οργανισμοί για καραντίνα. Αυτά λοιπόν επιτρέπουν τη συγκέντρωση στοιχείων ε, και ε, την ε, ενεργό δράση. Εξάλλου, αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων σε δεύτερο επίπεδο αυτό που ενδιαφέρει είναι στα σημεία εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ε, πρέπει να αποδίδουμε μεγαλύτερη προσοχή στις εισαγωγές να εντοπίζουμε τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν για συγκεκριμένα είδη φυτών. Τα μέτρα αυτά απαιτούν απαιτούν ε, δοκιμές ε, ή την εφαρμογή μιας περίοδου απομόνωσης ε, ή την απαγόρευση εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατά διάρκεια αυτού του διαστήματος πρέπει να γίνεται πλήρης αξιολόγηση των κινδύνων έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ληφθεί μία απόφαση είτε σε μόνιμη ε, βάση είτε με προσωρινά μέτρα. Επίσης ε, θέλω να σας αναφέρω ότι η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μικροβίων οργανισμών επιβλαβών οργανισμών μέσα, με τη μεταφορά στην Ένωση μέσα από τις αποσκευές των επιβατών αυτό ε, διαπιστώθηκε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ε, την εφαρμογή αυτού του καθεστώτος. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά στον κανονισμό είναι το βελτιωμένο και εξυγχρονισμένο πλαίσιο για το εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φυτά πρέπει να έχουν ένα διαβατήριο που τους ε, επιτρέπει τη μετακίνησή τους ε, στην επικράτεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα λοιπόν από αυτό το εναρμονισμένο και απλουστευμένο διαβατήριο φυτών προσφέρουμε την εγγύηση ότι τα φυτά και τα προϊόντα φυτών έχουν εξεταστεί ενδελεχώς και διαπιστώθηκε ότι δεν πρέπει να μπουν σε απομόνωση. Η απλούστευση και η εναρμόνιση ελέγχονται και κατά την έκδοση του διαβατηρίου και από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ως ε, συμβολή στις διαδικασίες ότι όταν τα φυτά πρέπει να συνοδεύονται με ένα ε, πιστοποιητικό πιστοποίησης ε, με βάση τους κανονισμούς για να πιστοποιείται η ποιότητά τους ε, τα δύο διαβατήρια, το, τα δύο έγγραφα με συγχωρείτε, το διαβατήριο των φυτών και η ε, ετικέτα πιστοποίηση, αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν. Επίσης, για να εκδοθεί το διαβατήριο ε, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταφύγει στην εποπτική αρχή. Το τρίτο στοιχείο του κανονισμού αφορά σε ένα βελτιωμένο σύστημα πιστοποίησης για εξαγωγές μέσα από την ε, πρόβλεψη ενός ε, πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από τα κράτη-μέλη όταν προϊόντα φυτών φυτεύονται ή την χάνουν μεταποίησης. Ε, αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό ε, μπορεί να εκδοθεί από το κράτος μέλος ε, χωρίς σημαντική χρονική καθυστέρηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα τρία στοιχεία κατά κάποιον τρόπο ανακεφαλαιώνουν τα νέα στοιχεία του κανονισμού και πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερη προστασία ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το εμπόριο. Ε, αυτός ο κανισμός δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα άρθρο το οποίο περιλαμβάνεται στις ε, τελικές διατάξεις και το άρθρο αυτό ορίζει καλύτερα τον ε, κανονισμό και επιτρέπει την ε, συγχρηματοδότηση κυρίως για ε, τη νέα κατηγορία επιπλαβών οργανισμών που μπορούν να συνεπάγονται ζημιές για τους εμπορευόμενους. Εξάλλου αυτός ο κανονισμός αντικαθιστά τις προϋπάρχουσες οδηγίες τις τέσσερις συγκεκριμένα που αφορούσαν στον έλεγχο επιβλεβών οργανισμών για τις πατάτες. έχει εφαρμοστεί ε, για τρία, ή μάλλον θα εφαρμοστεί για τρία χρόνια και πρέπει ε, εντωμεταξύ να θεσπιστούν και άλλες συμπληρωματικέ διατάξεις για να ολοκληρωθεί το καθεστώς προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει τώρα το λόγο. Mr. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, πράγματι, ε, ο συνάδελφος που αναφέρατε είναι εδώ. Εγώ όμως θα μιλήσω και εγώ είμαι ο Γιάννης Καραμίτσιος. Εργάζομαι για την Γαμαδέλτα Σάνκο. Οι προτάσεις ε, για το αναπαραγωγικό υλικό είναι μια πρόταση η οποία κωδικοποιεί και αντικαθιστά τις υφιστάμενες 12 οδηγίες για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και είναι πολύ σημαντικό τομέα αυτός γιατί τον λόγο υλικό αντιμετωπίζεται ως ακρογωνίος λίθος της γεωργίας αλλά και της όλης αλυσίδας ε, τροφίμων. Ε, με τον όρο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εννοούμε οποιοδήποτε φυτό ε, πηγαίνει προς την, ε, το σκοπό της αναπαραγωγής άλλων φυτών. Καλύπτει λοιπόν η πρόταση αυτή ένα φάσμα που πιάνει από σπόρους μέχρι πλήρως ανεπτυγμένα δέντρα. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται η χρήση του σκοπή στην αναπαραγωγή άλλων φυτών. Γεωγραφικά ε, γεωργικά δίκη, ε, είδη, διακοσμητικά φυτά, φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και πολλά άλλα καλύπτονται. Ενώ στην τρέχουσα πρόταση έχουμε νέε απαιτήσει βελτιωμένε για τα είδη που καλύπτονταν από τις προηγούμενε οδηγίε, αλλά καλύπτει και κάθε είδο φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Ωστόσο, με λιγότερο αυστηρές, αλλά δηλαδή πιο βασικές απαιτήσει. Η πρόταση αυτή εισάγει αρκετούς ε, σημαντικούς νεοτερισμούς σε σχέση με το εφιστάμενο καθεστώς, εκ των οποίων ένας είναι ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη ευθύνη για τους επαγγελματικού φορείς. Επίσης, άγεται μεγαλύτερη ευελιξία και είναι λιγότερο αυστηρές οι απαιτήσει για το υλικό το οποίο εξυπηρετεί την βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους, τη συντήρηση αυτών. Μιλούμε ιδίως για το υλικό των απομονωμένων, εξειδικευμένων αγορών, niche markets, των εξειδικευμένων ε, αγορών και επίσης ε, στόχος είναι και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών για να εξασφαλιστεί η ανεσοτημό ανταγωνισμού. και επειδή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της επίσημου ελέγχους θα εξασφαλίσει και την ανάκτηση κόστους. Πάλι για να έχουμε πιο δίκαιο ανταγωνισμό. Κάποια σημεία τώρα που ίσως να είναι σημαντικά για εσάς που θα εξετάσετε αυτή την πρόταση θα κληθείτε άλλωστε να την επεξεργαστείτε και να ψηφίσετε από αυτής. Αυτός ο κανονισμός πρώτα απ' όλα μεταφέρει την ευθύνη ε, στον φορέα ε, εκμετάλλευση ό,τι αφορά την πιστοποίηση του υλικού παράγει και διαθέτει στην αγορά. Από εδώ και πέρα όλοι οι φορείς θα μπορούσαν να έχουν την άδεια να πιστοποιούν από μόνοι τους το υλικό εφόσον πληρούν βέβαια συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και σε περίπτωση που δεν θεωρούν ότι είναι αρμόδιοι, δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους, προς αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τις αρμόδιες αρχές να λάβουν την πιστοποίηση. Όπως και να έχει όμως αυτή η πιστοποίηση θα γίνεται υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής οι φορείς θα μπορούν να θέσουν στο εμπόριο πιστοποιημένο υλικό, δηλαδή υλικό που υπόκειται σε υψηλό της απαιτησύνθος ή πρότυπο υλικό, standard material. Όμως για να εφαρμοστούν οι συνήθεις ε, πρακτικές για κάποια υλικά ιδίω αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, θα είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση, όπω συμβαίνει μέχρι τώρα για τα γεωργικά είδη, τα περισσότερα γεωργικά είδη, γεωργικέ καλλιέργειε. Η πρόταση θα παρουσιάζει λοιπόν περισσότερε απαιτήσει για την επισήμανση, τη συσκευασία, την χνηλασιμότητα, τι παρτίδε του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και ούτω καθεξής. Για τα ε, σημαντικά είδη των 12 οδηγιών για είδη που δεν έχουν ακόμη καταγραφή, όπως τα διακοσμητικά φυτά και το υλικό που χρησιμοποιείται για αυτά, εκεί πλέον εισάγονται μόνο βασικές απαιτήσεις, όπως για την επισήμανση ή αναφορά στην ονομασία των ποικιλιών. Αυτές οι βασικές απαιτήσεις είναι σημαντικές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλογή του καταναλωτή, η οποία θα γίνεται με γνώσεως ώστε να υπάρχει πίστη, αξιοπιστία και ε, εμπιστοσύνη μάλλον στην αγορά η οποία θα έτσι κυκλοφορεί ένα υλικό. Έρχομαι τώρα στην ε, καταχώρηση των ποικιλιών, το registration. Είναι σημαντικό για την πληροφόρηση των καταναλωτών, για να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές, το υλικό που εντάσσεται στις καταγεγραμμένες, ε, στα καταγεγραμμένα είδη, τα σημαντικά αυτά είδη, να μπορεί να, τεθεί, να στο εμπόριο αν ανήκει σε μια καταγεγραμμένη, καταχωρημένη ποικίλια. Αυτό είναι σημαντικό για τους ε, επαγγελματίες του κλάδου, για τους αγρότες, για τη βιομηχανία. Να ξέρουν τι ποικιλία, τι υλικό χρησιμοποιούν. Η καταχώρηση των ποικιλιών θα υπάγεται στο λεγόμενο DUS test για την ε, σταθερότητα, την ομοιογένεια και τη διάκριση. Distinction, uniformity, stability και στο VCU επίσης, Value for Cultivation In Use. Ή ε, στο α, κλασικό γεωπονικό αυτό τεστ ή στο sustainable VCU, βιώσιμο VCU. Θα κρίνεται δηλαδή με βάση την ε, περιβαλλοντική του επίδοση, το υλικό. και αν είναι σημαντικό το είδος θα μπορεί να υποβάλλεται σε όλους τους έλεγχους βυσιγιού όπως γίνεται συνήθως με τις γεωργικές καλλιέργειες. Η καταχώρηση των ποικιλιών μπορεί να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, να ε, καταχωριστεί δηλαδή μία φορά σε ένα εθνικό μητρό ποικιλιών και αργότερα να διατίθεται ελεύθερα στο εμπόριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή όμως τώρα εισάγει και μια δεύτερη επιλογή οι παρασκευαστές θα μπορούν να καταχωρίζουν σε ένα ε, μητρό της Ένωσης απευθείας ε, το υλικό τους, αν υπάρχει ευρύτερο συμφέρον για την ε, ευρωπαϊκή αγορά σε αφορά αυτό το υλικό. Η πρόταση, όπως προανέφερα, εισάγει νεοτερισμούς νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την προστασία της βιοπικιλότητας, τη διατήρηση των γενετικών πόρων, και την πρόθεση μικρών επιχειρήσεων. Απαγορεύεται η παραγωγή, μάλλον εξαιρείται από τους κανόνες η παραγωγή για ιδιωτική χρήση. Οι κυπουροί θα μπορούν Οι ερασιτέχνες θα μπορούν να παράγουν το υλικό που θέλουν. Μόνο για τράπεζες γονιδίων και τη διατήρηση γενετικών πόρων ε, όταν παράγεται ένα υλικό δεν θα υποβάλλεται σε αυτούς τους ελέγχους. Επίσης, ε, χαλαρή θα είναι οι κανόνες για την ε, καταχώρηση παραδοσιακών ποικιλιών. Θα είναι και μειωμένα τα τέλη. Ενώ οι εταιρείε που δεν έχουν μεγάλη παραγωγή θα εξαιρούνται οποιασδήποτε οποιοδήποτε τέλους. Όμως οι υλικά τα οποία παράγονται από μικροεπιχειρήσεις και πηγαίνουν ε, στην, ε, σε εξειδικευμένε αγορές δεν θα υποβάλλονται στην υποχρεωτική καταχώρηση των ποικιλίων. Μετά, με κατεξοδότηση πράξης, θα εγκρίνουμε κανόνες για το ετερογενές, ανομοιογενές υλικό όπως το λέμε. Δηλαδή ένα υλικό το οποίο δεν ανοίξει σε κάποια ποικιλία, αλλά αφορά συγκεκριμένους ε, πληθυσμούς, ε, συγκεκριμένα στρώματα. και ε, εγχώριες, εγχώριες φυλές. Τέλος, δασικό αναπαραγωγικό υλικό. Συμπεριλαμβάνεται γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό εξορισμού μιλάμε για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, άρα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. και θα πρέπει να υπάγεται και στους οριζόντιους ε, διατάξεις των επίσημων ελέγχων. Έχουμε την οδηγία το δασικό αναπαραγωγικό υλικό και θα πρέπει αργά ή γρήγορα να τροποποιηθεί η οδηγία αυτή για να ε, αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της συνέχισης της Λισαβόνας. Αφού θα έπρεπε λοιπόν να γίνει το άλλος, γιατί να μην το κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας για να μειώσουμε και το διοικητικό άχθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον επόμενο εκπρόσωπο της Κομισιόν. Εσείς αποφασίζετε μεταξύ σας ποιος θα λάβει το λόγο. Θα μιλήσω για την πρόταση της Επιτροπής για τη νέα νομοθεσία περί της υγείας των ζώων που θα απλοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την νομοθεσία για την υγεία των ζώων και θα έχουμε ένα ενιαίο ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία κατά των ασθενειών των ζώων. Ο βασικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής, μάλιστα, είναι να εξαλείψει τις μεταδιδόμενες νόσους μεταξύ των ζώων ή μεταδιδόμενες από τα ζώα στους ανθρώπους. Η πρόταση ε, περιέχει κάποιες αρχές για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, για ασφαλείς ε, μεταφορές των ζώων και των ζωικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, για την είσοδο και τις εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋποθέσεις αυτές, οι όροι αυτοί είναι σήμερα κατακαιρματισμένοι και ανεβρίσκονται σε 40 νομοθετικές πράξεις είτε του Συμβουλίου είτε του Κοινοβουλίου. Οι νομικές αυτές, νομοθετικές αυτές πράξεις θα αντικατασταθούν από έναν καινούριο ε, κανονισμό, ο οποίος ε, θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τη συνθήκη της, της Λισαβόνας με ε, εφαρμοστικές κατεξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής που θα υλοποιούν τον κανονισμό αυτό. Η νέα πρόταση λοιπόν αποσκοπεί σε μία μείζωνα απλοποίηση του ισχύοντος νομικού η πρόταση ε, βασίζεται στην εμπειρία του, της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη ζωική υγεία και περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε το 2007 με το σύνθημα «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Η καινούργια νομοθεσία θα καλύψει όχι μόνο την ε, ζωική παραγωγή αλλά και τους επιβλαβείς οργανισμούς και τα άγρια ζώα. Δεν θα καλύπτει ωστόσο το ευζήν των ζώων και, την, και τα κτηνιατρικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από άλλη νομοθεσία. Ε, το πιο σημαντικά καινούργια στοιχεία που εισάγονται με την πρόταση της Κομισιόν αφορούν την κατηγοριοποίηση και την ιεράρχηση των ασθενειών υπό την έννοια ότι τα κριτήρια για να αποφασίσουμε αν μια ασθένεια έχει ευρωπαϊκή σημασία θα γίνουν πιο διαφανή και πιο σαφή και θα βασίζονται περισσότερο σε μια αξιολόγηση κινδύνου. Το νέο νομικό πλαίσιο θα δώσει μια βελτιωμένη νομική βάση για την ανταπόκρισή μας σε νέες αναδιόμενες ε, ασθένειες που δυστυχώς έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρόσφατα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πιο συστηματικό επίσης σύστημα εποπτείας και πρόληψης των ασθενειών για τη βελτίωση της ασφάλειας θα υπάρχει μια ομαλοποιημένη, κεντρικοποιημένη προσέγγιση στον ευαλωισμό, εμβολιασμό και τα εμβόλια. Θα υπάρξει σύγκληση με τα διεθνή πρότυπα για την υγεία των ζώων που εκδίδει ο, οργανισμός για την, ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. Επίσης, κάποιες βασικές προϋποθέσεις για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που εξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναμένουμε ότι η καινούργια νομοθεσία θα στηρίξει και τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γενικότερα, ε, ο κανονισμός εισαγάγει αρκετά στοιχεία για πρόσθετη ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προσαρμόζουν στις τοπικές τους συνθήκες τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των ασθενειών, πάντοτε όμως εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα. Αυτή η καινούργια πρόταση δεν θα φέρει μια επανάσταση, αλλά πρέπει να ειδωθεί ως εξέλιξη ενός ομαλά λειτουργούντος και δρεωμένου συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ε, και τώρα Πάμε στον επόμενο μιλητή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι θα έχετε συμφωνήσει μεταξύ σας τη σειρά που θα μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω την τέταρτη νομοθετική πράξη αυτού του πακέτου που είναι η επίσημη έλεγχη. Η επίσημη έλεγχη είναι λοιπόν οι δραστηριότητες ε, τις ε, οποίες αναπτύσσουν οι ε, αρχές των κρατών μελών ε, για να διαπιστωθεί η συμβατότητα με την νομοθεσία. Υπάρχει ο ισχύων κανονισμός ε, και στον... Μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχει μια ε, πληθώρα δραστηριοτήτων που ε, καλύπτει αναλύσεις, τεστ και ούτω καθεξής. Οι κανόνες που ισχύουν τώρα, όπως σας είπα, έχουν καθοριστεί, περιλαμβάνονται στον κανονισμό 82 του 2004 που έχει σχέση ε, στην επαλήθευση της ε, ταυτότητας της ταύτισης ε, των κανονισμών γενικότερα με όσους προϋπάρχουν και εδώ κατ' ουσίαν μιλάμε για εγγυήσει και απαιτήσει που ισχύουν για τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων, η αμεροληψία, η τήρηση των ε, συνθήκων υγιεινής και ούτω καθεξής. Επίσης καθορίζονται κανόνες που αφορούν στη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των αρμόδιων αρχών ε, στους κτηνιατρικούς ελέγχους, στους συνοριακούς ελέγχους και το σημαντικότερο όλων αυτά αφορούν και στη χρηματοδότηση. Σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τις ε, βασικές αλλαγές όπως αυτές ε, προτείνονται στην ε, ε, πρόταση που εξετάζουμε. Η πρώτη λοιπόν σημαντική αλλαγή είναι η επέκταση του εύρους. Είπαμε λοιπόν ότι τώρα υπάρχουν λίγοι τομείς ε, που καλύπτονται από τον κανισμό 82 κάθετος 2004 κυρίως το πολλαπλασιαστικό υλικό και οι σχετικοί κανόνες δεν καλύπτονται, που σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού 82 όταν επαληθεύουν την συμβατότητα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Άρα δηλαδή αυτή είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή. Ο νέος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους, ο κανονισμός αυτός θα καλύπτει όλα τα το, τα κεκτημένα που έχουμε σχετικά με την προστασία των φυτών. Καλύπτεται λοιπόν το αναπαραγωγικό και πολλαπλασιαστικό υλικό και ορισμένοι κανονισμοί που είναι διάσπαρτοι αυτοί μπαίνουν κάτω από, την, το μανδύα του νέου κανονισμού. Αυτό ισχύει ας πούμε για κάποιους κανόνες σχετικά με ζυζανιοκτώνα ε, και ισχύουν και για τους ε, ε, κανόνες ε, κτηνιατρικής. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν κάτω από το μανδύα του ίδιου ε, κανονισμού. Ας δούμε εκείνο που απομένει. Απομένει μια βασική αρχή σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που λέει ότι θα πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος. Οι αρμόδιες αρχές ε, διεξάγουν ε, εποπτικές ε, δραστηριότητες αξιολογώντας τον κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τον αντικειμενικό κίνδυνο, τον εγγενή κίνδυνο σε διάφορες περιοχές, διεξάγουν λοιπόν ελέγχους, αυτά παραμένουν. Εκείνο που είναι νέο και προστίθεται είναι ότι εκτός από αυτούς τους ε, ελέγχους ε, που περιλαμβάνονται στο πολιετές ε, πρόγραμμα ελέγχου το οποίο καλύτερα να καταρτίζει κάθε αρμόδια αρχή, τα κράτη-μέλη καλούνται σε αυτά τα προγράμματα να περιλαμβάνουν και κανονισμούς κατά της απάτης. Δηλαδή, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία, αλλά σε συγκεκριμένες δραστηριότητε αντιμετωπίζεται ε, η απάτη, η παραβίαση με δόλο. Οι έλεγχοι ε, είναι ξαφνικοί, χωρίς να έχουν ε, ανακοινωθεί και επειδή τελικά έχουμε συνοψίσει όλους τους κανόνες περί ελέγχων, έχουμε διαγράψει κάποιες άλλες πράξεις οι οποίες διέπουν αυτή τη στιγμή τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών και προσφέρουμε μία σειρά διατάξεων έτσι ώστε να επιτρέπεται η θέσπιση ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι βασικές διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στους νέους ελέγχους θα μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τομέα. Στη νέα λοιπόν πρόταση προβλέπεται προβλέπονται εξουσιοδοτήσεις για συγκεκριμένους ε, ελέγχους, ε, παραδείγματος για τους ελέγχους ε, σε μεταλλαγμένα προϊόντα ή ελέγχους που έχουν σχέση με την ευημερία των ζώων. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί τομείς όπου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή των βασικών κανόνων στις ανάγκες του κάθε τομέα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι για να εγκριθούν νέες απαιτήσει, νέοι έλεγχοι, σε, αν προκύψει κάποιος καινούριος κίνδυνος, εκεί αυτά προκύπτουν με βάση ε, νέα μοντέλα κατανάλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο κανονισμός δεν προβλέπει ειδικέ ε, διατάξεις περί ελέγχων. Ε, εδώ προβλέπεται μόνο ότι ισχύουν οι κατεξοδότηση πράξης. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο του κανονισμού περί ελέγχων είναι το κεφάλαιο σχετικά με τη διοικητική αρρωγή και τη συνεργασία. Μία από τις δυσκολίες ε, για την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι αρμόδιες αρχές δεν εξαντλούν τις προνομίες και τις δυνατότητες που έχουν να συνεργάζονται ε, με τους ε, συναδέλφους τους σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν που προτείνεται να πράξει πρόταση είναι να ενισχύσει την διοικητική αυτή αρρωγή σε όλες τις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία και πέρα από τα σύνορα. Αυτό ισχύει για κάθε μορφής ε, παραβιάσης συμπεριλαμβανομένης και της απάτης. Στην πρόταση θα περιλαμβάνονται αυστηρές ημερομηνίε, υποχρέωση ανταπόκρισης. Πρέπει επίσης να βελτιωθούν τα εργαλεία ε, μέσα από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει την διασυνοριακή διοικητική αρρωγή. Τα εργαλεία που υπάρχουν για το σύστημα ελέγχου οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επωφεληθούν από την ε, χρησιμοποίηση διαφόρων εργαλείων πληροφορικής που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, τα κρατημέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεργάζονται. Κάτι που είναι γνωστό είναι το σύστημα ταχείας προειδοποίησης ε, για τα τρόφιμα, αλλά υπάρχει και άλλο σύστημα ε, πληροφορικής, ε, το Eurofeed, το Tracy System. Υπάρχουν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στο νέο σύστημα ελέγχων. Επειδή μιλάμε για τα εργαλεία και τα μέτρα, ε, αναφέρθηκε ήδη στην πρώτη παρέμβαση ότι ε, θα προβλέπονται νέες ε, κυρώσεις σε περίπτωση απάτης, διότι οι διατάξεις περί της, του αποτρεπτικού στοιχείου των κυρώσεων προϋποθέτει ότι οι χρηματικές, τα χρηματικά πρόστιμα θα πρέπει να είναι τέτοιου ύψους έτσι ώστε ε, να μην προκύπτει οικονομικό όφελος από την παραβίαση. Να υπάρχει δηλαδή σαφώς αποτρεπτικός χαρακτήρας της ε, κύρωσης. Μία άλλη σημαντική καινοτομία αφορά στην συμπερίληψη των διαφόρων ελέγχων στα σύνορα. Αυτά όλα εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα με κοινούς μηχανισμούς, κοινά έγγραφα και κοινά σημεία εισόδου. Που σημαίνει ότι τα διάφορα καθεστώτα ελέγχου συνόρων που ισχύουν για τα κτηνιατρικά προϊόντα, ε, για τα ε, φυτά και για άλλα προϊόντα μη ζωικής προέλευσης. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα έτσι ώστε οι εμπορευόμενοι να μπορούν να έχουν έναν ενιαίο κανονισμό ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εμπορίας που ελέγχεται στα σύνορα. το που τράβηξε ενδιαφέρον είναι η χρηματοδότηση των ελέγχων. Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι η εξή. Ορισμένα τμήματα της αλυσίδας τροφίμων πληρώνουν για τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Ας πούμε ένα σφαγείο πληρώνει για τους συνεχείς ελέγχους από τις αρμόδιες εκτινετρικές αρχές. Αυτό όμως δεν ισχύει για άλλους ε, τομείς. Αυτό ισχύει μόνο για κάποιους, ε, για αυτούς που παράγουν άλευρα, ε, ψάρια, ασχολούνται με την αλεία. Τώρα η νέα πρόταση προβλέπει την υποχρέωση, των κρατών μελών να χρηματοδοτούν μόνες, μόνα τους τα κράτη-μέλη τους ελέγχους. Άρα πρέπει να έχουν οικονομικά αποθέματα για να εφαρμόζουν την νομοθεσία και προβλέπονται και ε, υποχρεωτικά τέλη. Δηλαδή επιβάλλονται τέλη σε όλους τους εμπορευόμενους που υφίστανται ελέγχους ε, της, από την αλυσίδα ή που εμπορεύονται προϊόντα της αλυσίδας τροφίμων. Αυτό νομίζω ε, έχει αναφερθεί. Ε, μόνη σημαντική εξαίρεση είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές δεν θα πληρώνουν. Και αυτές βέβαια θα ελέγχονται ανάλογα με τον κίνδυνο που προκαλούν, αλλά δεν θα καλούνται να πληρώνουν για τους ε, ελέγχους που θα υφίστανται. Αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό βάρος ε, θα μετακυλείται στους άλλους εμπορευόμενους της αλυσίδας. Ο κανονισμός λέει βέβαια ότι δεν πρέπει να υπερβάλλονται υπερβολικά οι υπόλοιποι επειδή δεν πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε γενικές λοιπόν γραμμές θέλω να πω ότι διευρύνεται η εμβέλεια για να καλύπτεται το σύνολο της αλυσίδας ε, τροφίμων και επιβάλλονται τέλη τα οποία προβλέπεται να καλύπτουν ε, το κόστος ε, που απορρέει από τους ελέγχους. Οι εμπορευόμενοι λοιπόν πλήρους απασχόλησης ε, καλούνται να πληρώνουν, όμως αυτοί θα επωφεληθούν και από τις προτινόμενες αλλαγές, διότι η πρόταση βελτιώνει τη διαφάνεια του συστήματος, άρα δηλαδή οι μεταποιητές τροφίμων θα πρέπει να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να επιβάλλουν τα τέλη. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και αυτοί επίσης θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το πώς καθορίζονται τα τέλη και πώς επιμερίζεται το κόστος ε, στους διάφορους τομείς και στα διάφορα τμήματα της αλυσίδας. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στις ε, πληροφορίες ε, και στις ε, ρυθμίσεις που προτίθεται να επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την επιβολή τελών να ε, δαπανώνται λογικά, ορθολογικά αν θέλετε. Αυτές είναι οι ε, διαφανείς διατάξεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση σχετικά με τη συγκέντρωση των χρημάτων και πώς αυτά δαπανώνται. Γενικότερα τώρα για τη διαφάνεια αυτή δεν έχει σχέση μόνο με μεθόδους για τη χρηματοδότηση των ελέγχων, αλλά έχει σχέση γενικότερα με την πρόσβαση που αποκτούν οι πολίτες, που μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι αρμόδιες αρχές ε, εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους εφαρμογή ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων. Η πρόταση ενισχύει τις απαιτήσει διαφάνειας, απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να ε, δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για ελέγχους, για ευρήματα, ε, για ε, μη συμβατότητα, για ενέργειες που αναλαμβάνονται σε περίπτωση μη συμβατότητας, άρα δηλαδή ε, οι αρμόδιες αρχές προληπτικά δημοσιεύουν πληροφορίες και επιπρόσθετα οι αρμόδιες αρχές με μεγαλύτερη ευκολία δίνουν τη δυνατότητα διάδοσης πληροφοριών για τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων σε ε, συγκεκριμένους εμπορευόμενους. Επίσης ε, δίνουν τη δυνατότητα ευκολότερα μπορεί κανεί να καταφύγει σε προγράμματα βαθμολόγηση, δηλαδή προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα σε πολίτες να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των ελέγχων. Βλέπουν ε, πως ε, τη βαθμολογία συγκέντρωσε ένας ε, λιανέμπορος ή ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια του ελέγχου και από εκεί βεβαίω ρυθμίζουν και την αποφασή τους σχετικά με το τι θα καταναλώσουν. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι, δύο λόγια κύριε Πρόεδρε για να ολοκληρώνουμε. Θα συνοψίσω. Είδατε ότι οι τέσσερις αυτές προτάσεις αποτελούν ένα τεράστιο πακέτο που θα έχει αποτέλεσμα την ε, πλήρη αναθεώρηση ομοθεσίας ε, για τα τρόφιμα, την τροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Θα εξορθολογήσει όλη την νομοθεσία, θα καταργήσει πάρα πολλέ νομοθετικέ πράξει που ήσχαν μέχρι τώρα. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ε, βέβαια αν δεν υπάρξει και η υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την οικονομική. Εγώ μίλησα και για κάποιες προτάσεις. Η πέμπτη πρόταση που έχει καθυστερήσει μάλλον θα εγκριθεί από την Κομισιόν στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Με αυτή την τελευταία πρόταση λοιπόν που επαναλαμβάνω θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα θα έχετε κι εσείς στη διάθεσή σας το πλήρες πακέτο για να αποφασίσετε πού πηγαίνουμε με τη γεωργία, με τη τροφική αλυσίδα από σπόρους, ε, φυτά ζώα και τις προτάσεις που έχετε επιτάπητος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στις 13 Ιουνίου διοργανώνουμε μία διάσκεψη. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και ευπρόσδεκτοι οι ευρωβουλευτές φυσικά, όπου θα εξηγήσουμε αυτές τις πέντε προτάσεις ε, πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας συνοψίσατε τις παρουσιάσεις που ακούσαμε πληρέστατες παρουσιάσεις, αναλυτικότατες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. και ζητώ συγγνώμη που δεν σας ε, παρουσίαζα με το ονοματεπώνυμό σας, αλλά δεν είχα ε, στη διάθεσή μου τη σειρά με την οποία θα παίρνετε το λόγο. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Έχω επτά εγγεγραμμένους. Κυρία Γέγκλη είναι η πρώτη ομιλήτρια. Και σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Θα σας ε, ενημερώνω όταν πλησιάζει να εκπνεύσει ο χρόνος σας. Τρία λεπτά ο καθένας λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό το ότι οι βουλευτές έχουν λιγότερο χρόνο να παρεμβαίνουν από τους υπόλοιπους. Αυτά που ακούσαμε πραγματικά ήταν πάρα πολύ λεπτομερή. Τώρα τα συζητάμε όλα χίδιν, φίρδιν, μίγδιν. Εγώ ε, ήθελα να μιλήσω γενικότερα για την ε, υγεία των ζώων και λυπάμαι που μόλις μιλήσω θα αναγκαστώ και να φύγω γιατί δεν υπολογίζω ότι θα μιλήσει τόση πολύ ώρα η Επιτροπή. Κοιτάξτε, καταρχήν να ευχαριστήσω και να πω ότι εδώ και πολύ καιρό περιμέναμε αυτές τις ε, προτάσεις. Να πω όμως και το εξής και θα το πω με απόλυτη σαφήνεια. Από την πρώτη πρόταση που ακούσαμε μέχρι και την τελευταία γίνεται λόγος για μεταρρύθμιση. Και θέλω να σας πω, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρέθηκαν, κουράστηκαν να ακούνε συνέχεια για μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε τι θέλουν, θέλουν βελτιώσεις, απλουστεύσεις. Εντάξει, το είπαν και αυτό οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, αλλά βλέποντας γενικότερα ε, το τι προκύπτει δεν βλέπω να υπάρχουν και πολλές απλουστεύσεις, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Είναι σωστό πράγματι να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Στον τομέα της ε, υγείας και της προστασίας των ζώων έχουμε ζητήσει επανειλημμένα απαρχαιωμένες προτάσεις επιτέλους να τις εξυγχρονίσουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν λοιπόν μεμονωμένα σημεία που είναι σημαντικά που αφορούν σε ασθένειες ζώων, που αφορούν ε, στη μετάδοση των ασθενειών. Γίνεται σε επανειλημμένα για την εισαγωγή ζώων και ζωικών ε, προϊόντων, αλλά δεν ελέγχθη τίποτα για τις εξαγωγές. Και σε σχέση με τις εξαγωγές ε, δεν γίνεται και πολύ λόγος για τη μεταφορά των ζώων, που θα είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Επίσης, ε, ελέγχθη ότι οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στην κοινή αγορά, αλλά να μην ε, αγνοούν το, την ιδιομορφία των ε, περιφερειών. Εμείς ε, την ιδιομορφία θέλουμε να τη διατηρήσουμε την ιδιομορφία των περιφερειών για όλα τα προϊόντα και να μην επιτύχουμε, να μην οδηγήσουμε σε ισοπαίδωση των προδιαγραφών στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Τελικά, όταν θα τα διαβάσουμε όλα αυτά, με ενδιαφέρει να δω πώς θα είναι αυτό το βελτιωμένο πλαίσιο και πώς ε, θα γίνονται αυτοί οι βελτιωμένοι έλεγχοι. Σε όλες τις ε, εκθέσεις ε, αναζητάται ο κοινός παρανομαστής ανάμεσα στην κοινωνία, την γεωργία, τον καταναλωτή. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλα τα σημεία που παίζουν ρόλο και σας το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Δεν πρέπει να στυλιτεύουμε τη γεωργία, πρέπει να εξετάζουμε το σύνολο της αλυσίδας το κάναμε αυτό και με το αλογίσιο κρέας ε, που δεν είχε καμία σχέση με την ε, γεωργική παραγωγή αλλά με άλλου είδους θέματα. Η χνηλασιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ε, συμφωνώ επ' αυτής, αλλά όπως σας είπα, τους ε, μεταποιητές ε, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως συμμάχους μας και τους καταναλωτές και δεν πρέπει απαραίτητα να τα με μεταρρυθμίσεις απλά να βελτιώσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ταραμπέλα, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Αυτά τα τρία πολύ σημαντικά σημεία διάταξη. σίγουρα πρέπει να τα συζητήσουμε και ίσως να αποτελέσουν και αντικείμενο μια ακρόασης ε, γιατί όπως είπαν και εκπρόσωποι πολύ μεγάλος αριθμός 80 νομοθετικές ε, πράξεις ε, θα καταργηθούν ε, με, αυτό το, ε, με αυτές τις νέες πέντε προτάσεις. Θέλουμε λοιπόν να, να υιοθετώσουμε αυτούς τους νέους κανόνες που θα συγκεντρώνουν 12 οδηγίες. Από το 66 είναι ο πρόσφατος και πραγματικά θέλουμε να φροντίσουμε και τη βιοπικιλότητα. Ξέρουμε ότι 75% ε, έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Επίσης, 10 μεγάλες επιχειρήσεις ε, στο παγκόσμιο επίπεδο έχουν τα 3 τέταρτα ε, των σπόρων που χρησιμοποιούνται. Δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε ταυτό εξού και είναι σημαντικό και να κάνουμε τη διατύπωση πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση και να προστατεύσουμε τις ποικιλίε ε, και αυτό περισσότερο από ποτέ όταν λέω τις προστατεύσουμε χωρίς όμως να επιβάλλουμε, να επιβάλλουμε πολλούς περιορισμούς. Φοβούμε λοιπόν ότι ναι μεν υπάρχουν χαλαρώσεις, κατάλαβα πολύ καλά τι είπε της Κομισιόν, προβλέπονται χαλαρώσεις κάποιων απαιτήσεων σε ό,τι αφορά την καταχώρηση, το registration, αλλά ε, επειδή είχα καταθέσει μια ερώτηση τον Ιούλιο πέρυσι και απάντηση κομισιών για μια πιο ελαφρυμένη διαδικασία για τους πόρους που χρησιμοποιούνται, τις διαφορετικές ποικιλίε που χρησιμοποιούνται. Εγώ ε, μπορεί να μην είμαι μέλος της Ένωσης, αλλά ε, υπάρχει μια ένωση, η λεγόμενη Κοκοπελή, που το εφετείο του Νανσί την καταδίκασε μετά από προδικαστικό ερώτημα που είχε θέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ό,τι αφορά του σπόρου που δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο. Υπάρχουν λοιπόν ελαφρύνσει πράγματι σήμερα, αλλά ακόμα είναι βαριέ οι απαιτήσει. 580 ε, ε, είναι οι περιπτώσεις οποίες είχαμε ελάφρυνση μόνο. Άρα πρέπει να απελευθερώσουμε κάπως τα πράγματα. Ε, να πλουστεύσουμε την κατάσταση, ώστε πράγματι ένας αρασιτέχνης ε, κυπουρός, ε, ο κυπουρός της Κυριακής και άλλοι μικροί παραγωγοί να μπορούν με κάθε ελευθερία και στο μέλλον να συνεχίσουν τη δραστηριότητα, δεν απειλούν αυτή την υγεία των πολιτών. Δεν μπορούμε να του ταυτίσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτά πρέπει λοιπόν να τα επιτρέψει ο νέος κανονισμός. Δεύτερο τώρα, και έρχομαι προς τη γάμα Δέλτα Άγκρη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισαμε ένα τέρας στο Στρασβούργο. Ψηφίσαμε ένα ψήφισμα που ανοίγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Μια τεράστια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα. Γιατί το λέω τέρα, όχι ότι δεν πρέπει να δερματευτούμε με τον άλλο μεγάλο παγκόσμιο πρωταγωνιστή σε οικονομικά θέματα, αλλά πώ λάβαμε την απόφαση. Πώς περάσαμε αυτό το ψήφισμα, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες. Ε, δεν νομίζω ότι θα το κάνει η αρμόδια γάμα δέλτα της Κομισιόν. Γι' αυτό στρέφω στη γάμα δέλτα αγκρή, γιατί ε, υπάρχει αυτή η πολιτιστική εξαίρεση. Καλά κάναμε, αλλά δεν μιλήσαμε αρκετά για την προστασία, για τα ζωτούχα, για τα φυτοφάρμακα, η οδηγία REACH ε, για τα χημικά ε, μόρια, τα πλανητικά κτλ, κτλ. Αν ξεκινήσουμε συνομιλίες και δεν μιλήσουμε για ένα κίνδυνο, την αμοιβαία αναγνώριση για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει ε, η Κομισιόν να, να αντισταθεί. Δεν ξέρω ποιος επίτροπος, μπορεί να είναι και ο ίδιος, πάντως αρμόδιος για τη Γεωργία Επίτροπο. Πρέπει να κάνει τι κινήσει του ο έλεγχο επίση, και αυτό που είπε η κυρία, ναι, συμφωνώ. Αλλά αν έχουμε ένα μηχανισμό ελέγχων που τελικά εκ των υστέρων δούμε ότι αφού δεν έχουμε κάνει τι διαπραγματεύσει μα ε, σε ό,τι αφορά την ΕΜΒΕ αναγνώριση, δεν τον κάνουν τον έλεγχο μετά. Και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Οι Αμερικανοί που είναι πάρα πολύ ρεαλιστές και ικανοί προσπίζονται συμφέροντά τους και εμείς ανοίγουμε την πόρτα πολύ περισσότερο ουσιαστικά ανοίγουμε την πόρτα στην ε, απόρριψη των κανόνων που εμείς θέλουμε να ισχύουν. Και ε, θα φτάσουμε σε επιβλαβείς ε, εξελίξεις για το γεωργικό τομέα αν περάσει αυτό το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πόλσεν έχει τώρα το λόγο θα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση. Και υπάρχει μπροστά μας μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Ε, εισηγήτρια πριν από 10 χρόνια ε, για τον κανονισμό περί των ελέγχων και οφείλω να πω ότι έχω παρακολουθήσει τον ε, κανονισμό αυτό στην ηλική του εφαρμογή επί 10 χρόνια. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλω να πω στον εισηγητή του Κοινοβουλίου. Καταρχήν η ανάλυση κινδύνου. Στην πραγματικότητα αυτή η ανάλυση λειτουργεί πάρα πολύ άσχημα. Γιατί? Γιατί η πλειοψηφία των, των υπεύθυνων των ελέγχων προτιμούν να βάζουν ό, τα πάντα στην κατηγορία επικίνδυνο ή πολύ επικίνδυνο. Ε, πράγμα που προκαλεί και δημιουργεί πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και προβληματισμό ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω Το σύστημα των ε, δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ε, των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ περίπλοκο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πια μικρά σφαγεία στην Ευρώπη. Άρα η μεταφορά ζωντανών ζώων διαρκεί πολύ περισσότερο και διανύει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνεκτική στάση. Όσο αφορά τώρα την έκθεση για την υγεία των ζώων, πρόκειται για ένα θέμα που γνωρίζω πολύ καλά. ε, ίσως όχι μέχρι και την τελευταία τεχνική πτυχή του θέματος, αλλά ε, η ελεύθερη ανταλλαγή, συμφωνία ε, σε ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή, με την Συναμένες Πολιτείες, εσωτερική αγορά κτλ. κτλ. Είμαι φιλελεύθερη, είμαι πεπισμένη ότι η ελευθερία των συναλλαγών είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν θέλω μια ελεύθερη ανταλλαγή ασθενειών, για παράδειγμα. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία. Από τη μία πλευρά πρέπει να προστατευθούμε από τους κινδύνους ε, και βεβαίως υπάρχει και η ελευθερία των συναλλαγών. το σύνδεσμο μεταξύ της υγείας των ζώων και της υγείας των ανθρώπων και με ανησυχεί πάρα πάρα πάρα πολύ η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ε, πρέπει εδώ να βρούμε τον κρίκο, τη σύνδεση. Ε, όταν θα μπούμε στις λεπτομέρειες θα σας ζητήσω να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι στην διατροφική ε, αλυσίδα υπάρχουν ακριβώς αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν πρέπει να χανόμαστε στις λεπτομέρειες, αλλά να έχουμε μια συνολική όψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Έχει τώρα το λόγο και μετά κυρία Ράιμερς. Κύριε Πρόεδρε, είναι βεβαίω ε, πάρα πολύ δύσκολο μετά από αυτού του ατέλειωτου μονολόγου Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει κανεί σε τρία μόνο λεπτά για τόσο σημαντικά θέματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ε, ή θα έπρεπε ε, να έχουμε περισσότερο χρόνο ή να μοιράσουμε τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ, εν περιπτώσει, τώρα θα περιστώ στο θέμα των σπόρων, διότι είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις που θα κατατεθούν και θα σκηθεί δρυμύτατη κριτική για αυτά που έχουν προταθεί. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κουνήθηκε, αλλά θα πρέπει να μου εξηγήσουν γιατί τώρα βάζουν το όριο στα 2 εκατομμύρια κύκλο εργασιών ε, στους 10 συνεργάτες. Πώς, πώς ορίστηκε αυτό το ανώτατο όριο. Ή μας, ξέρετε μας πείτε γιατί τα 2 εκατομμύρια είναι το όριο και μετά αυτό το περίφημο νίσο, αυτή η σφήνα, τι σημαίνει, ε, τι σημαίνει για πολλούς. Ε, ε, Μπορεί κανείς να πουλάει μόνο σε περιφερειακές αγορές ή σε τοπικές αγορές. Η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει εδώ πολύ έξυπνα τρίκ και τι λέει στο τέλος, ξέρετε τα υπόλοιπα θα ρυθμιστούν με κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτό όμως δεν βοηθάει, δεν βοηθάει να επιτύχουμε το στόχο μας ούτε και της Επιτροπής. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η Κομισιόν πώς αντιδρά στο ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ουσιαστική μείωση των μονάδων καλλιέργειας και των ποικιλιών. Και πώς εντάσσονται αυτά στην στρατηγική βιοπικιλότητας. Δηλαδή πρέπει κανείς να το δει το θέμα και από την άλλη πλευρά. Δεν μας ενδιαφέρει ο συγκεντρωτισμός, αλλά η ποικιλομορφία. Και δεν βλέπω να υπάρχει. Πού είναι η στρατηγική εκείνη που εμποδίζει όλο και περισσότερες εταιρείες να οθούνται, να σπρώχνονται σε μία αγορά, ε, κυρίως ε, χημικές εταιρείες. Δεν πρόκειται μόνο για, την, ε, για τις οικολογικές καλλιέργειες, πρόκειται και για πολλές τοπικές καλλιέργειες που δεν είναι δυνατόν όλοι οι σπόροι να καταλήγουν σε τράπεζες σπόρων. Εγώ δεν το βρίσκω καλό να γίνονται καλλιέργειες για να καταλήγουν οι σπόροι ε, σε ειδικέ ε, τράπεζες. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. Ε, υπήρχε μια πεπατημένη και πρέπει αυτή να συνεχιστεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφωνώ με αυτό που λέγεται ότι για να διατηρηθούν οι ποικιλίε θα πρέπει να καταφύγουμε στις τράπεζες γονιδίων. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. Το ερώτημα λοιπόν που με απασχολεί είναι το εξής. Σε τελική ανάλυση πώς μπορούμε να εμποδίσουμε κυρίως τον τομέα των ε, κυπευτικών να προκύπτει αυτή η υπερβολική τάση προς ε, βρυδιακές καλλιέργειες. Δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι σπόροι αλλά τα υβρίδια. Εγώ αυτό το κατακρίνω. Και σε τελική ανάλυση αφαιρούνται δυνατότητες επιλογής από τον καταναλωτή. Σε αυτά τα θέματα δεν βλέπω να έχει δώσει απαντήσει η Κομισιόν. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τις καλές τους προθέσεις. εντάξει, πιστεύω ότι ήθελαν πολλούς κανονισμούς να τους συγχωνεύσουν σε έναν και μόνο ή σε λιγότερους. Αλλά παρόλα αυτά τίτε το ερώτημα ε, σε αυτό, αυτή την προσπάθεια του συγκεντρωτισμού δεν θυσιάζουμε την ποικιλομορφία και έχετε δει και μόνοι σας πώς αντιδρά η κοινή γνώμη σε τέτοιου είδους ε, προτάσεις. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι αυτοί οι κανονισμοί τελικά εκφυλίζονται. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να επιτύχουμε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι συγκεντρωτισμό, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, με το συγκεντρωτισμό χάνεται η περιφερειακή ποικιλομορφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω ότι Τώρα ξεκινάει όλη η διαδικασία, τώρα ξεκινάνε οι εργασίες, άρα θα έχετε πολύ χρόνο και πολλές ευκαιρίες να πάρετε το λόγο. Και μετά Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν, ε, όσον αφορά τους επιβλαβείς ε, οργανισμούς. Μέχρι τώρα τι γινόταν. Οποτεδήποτε εμφανιζόταν ένας τέτοιο επιβλαβής οργανισμός, οι εταιρείε που το δήλωναν ήταν και αυτές που τιμωρούνταν. Γιατί, γιατί έπρεπε να καλύψουν μόνες τους ε, τη ζημιά του. Μήπως λοιπόν ε, να πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα έτσι ώστε οι εταιρείε που εντοπίζουν αυτή την ε, διείσδυση των επιβλαβών οργανισμών να μην τιμωρούνται. Όσον αφορά ε, τον πολλαπλασιασμό φυτών πρέπει να έχουμε υπόψη. Όταν πρόκειται για φυτά δασοκομείας, εκεί το σύστημα πολλαπλασιασμού είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στη Γεωργία. Δηλαδή, ε, πρέπει να μαζευτούν οι σπόροι και μετά να πολλαπλασιαστούν σε ειδικέ εγκαταστάσεις ε, σε τελείως, με τελείως διαφορετικές συνθήκες ε, από ό,τι στη Γεωργία. Ε, στη Γεωργία, όπως σας είπα, είναι άλλες συνθήκες, άρα δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα και η διομορφία της δασοκομεία πρέπει να διατηρηθεί. Όσον αφορά την υγεία των ζώων, πράγματι χρειαζόμαστε αποτελεσματική προστασία από μολυσματικές ασθένειες στην Ευρώπη από επιδημίες. Επίσης, ε, οι ασθένειες, οι μολυσματικές ε, ε, που μεταδίδονται με τα κουνούπια αυτές οδηγούν σε εμπορικούς περισμούς που βλάπτουν όλο τον τομέα. Δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε τα κουνούπια να έρχονται στην Ευρώπη. Πρέπει όμως οι ε, κτηνοτρόφοι να ξέρουν ότι δεν θα καλούνται μόνοι τους να καλύψουν τη ζημιά. Όσον αφορά τους ελέγχους πρέπει να είναι σαφές ότι έχουμε διαφορετικά κρατικά συστήματα. Έχουμε συστήματα έντονα κρατικά στα κρατημέλη και άλλα ομοσπονδιακά, περιφερειακά. Εάν λοιπόν θέλουμε την ομοιομορφία πρέπει να έχουμε κατά νου το ένα σύστημα να μην βλάψει το άλλο. Πρέπει να εξευρεθεί ένας ε, τρόπος για να μπορούμε να προσαρμόσουμε και τους ελέγχους. Κατόπιν είπατε ότι στο μέλλον το κόστος θα καλύπτεται από την επιβολή τελών και πρέπει να προσέξουμε, διότι όταν επιβάλλουμε ε, τέλη ε, ενδέχεται να δημιουργηθεί μια λυσίδα όπου τελικά θα πληρώνει ο τελευταίος κρίκος. Δηλαδή, πληρώνει το σφαγείο και τελικά, ποιος τραβάει όμως ε, την όλη υπόθεση, είναι ο απλός κτηνοτρόφος, ο πιο αδύναμος κρίκος. Γιατί στην περίπτωση αυτή, αντί να επιτύχουμε το στόχο μας, απλά επιτείνουμε το πρόβλημα. Το βρίσκω πάρα πολύ συμπαθητικό το ότι μας καλείτε ε, στην συνδιάσκεψη αυτή ε, για τα θέματά σας. Ε, είναι όμως μια ημερομηνία που πέφτει στην Ολομέλεια Στρασβούργου. Αυτό για μας δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έρθουμε, δεν μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Ίσως θα ήταν συμπαθητικό η Κομισιόν να έχει κατά νου τις εβδομάδες του Στρασβούργου και να μην συζητάει τόσο σημαντικά θέματα χωρίς εμάς. Αυτά πολύ σύντομα. Δεν, δεν είχαμε χρόνο ε, να απαντήσουμε. Καλό που αναφερθήκατε σε τόσες λεπτομέρειες, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ελπίζω αυτό να διορθωθεί στο μέλλον. będzie taka szansa zapewne. E, ο κύριος Σιλβέστρης και μετά κύριε Παλάτσο. Ευχαριστώ. Όχι, ο κύριος Σιλβέστρης πρώτα, μετά εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου και τη συμφωνία μου με αυτήν την ιδέα ενός πακέτου τεσσάρων προτάσεων προς το Κοινοβούλιο που είναι απαραίτητες για την εδραίωση και την καλύτερη ενοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πλήρως με την ανάγκη να φέρουμε σε ένα ενιαίο κείμενο ε, ιδίως τα όσα αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό ε, υλικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο 12 διαφορετικών οδηγιών. Ε, πρόκειται για ένα κείμενο ε, στο οποίο πρέπει να βρούμε κάποια σταθερά και συμφωνημένα σημεία ισορροπίας. Ε, συμμερίζομαι όσα είπε ο συνάδελφος Ταραμπέλα στην ε, εισήγησή του. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι σημαντικά και πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ πολλών απαιτήσεων. Είναι η απέτηση της λασιμότητας, θεμελιώδους σημασίας, μία από τις αρχές της θεμελιώδης αυτού του εγγράφου. Υπάρχει ανάγκη ε, πρόληψης επίσης, ανάγκη Πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων. Η χνηλασιμότητα γι' αυτό ε, είναι θεμελιώδης. Ε, πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σταθερότητα του υλικού. Πρέπει να υπάρχει επίσης ο έλεγχος στην εμπορευματοποίηση των σπόρων και εκεί επισέρχεται η χνηλασιμότητα. Υπάρχει ανάγκη να εγγυηθούμε στις μικρές επιχειρήσεις ή στους μικρούς καλλιεργητές. Ένα όριο στην ε, εμπορική τους δραστηριότητα για να, ε, ε, και να αποφύγουμε ένα πρόσθετο, μια πρόσθετη γραφειοκρατία που θα επιφέρει κι άλλο κόστος. Νομίζω ότι η δουλειά που μας περιμένει και που θα είναι πολύ εντατική ε, και αφήνω κατά μέρος τη, τις δυσκολίες, την πρόληψη, την αποσαφήνιση, τη διασαφήνιση, τη λιγότερη γραφειοκρατία, τη βοήθεια προς τις αγορές για τη διάθεση των προϊόντων πάνω από όλα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια σημεία ισορροπίας πάνω στα οποία παίζεται ακριβώς ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, πέρα από, την, ε, από το να εγγυόμεθα τη δραστηριότητα των μεγάλων εταιριών χωρίς όμως να ποινικοποιούμε και να περιθωριοποιούμε τους μικροκαλλιεργητές. Όλα αυτά έχουν βέβαια και ένα κόστος, πάνω στο οποίο πρέπει να παρέμβουμε έντονα. Μιλά, γίνεται λόγος για ευελιξία και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε και να εργαστούμε. Όπως είπα, επισήμανση η χνηλασιμότητα, ε, τομείς στους οποίους πρέπει να δράσουμε με τη μέγιστη προσοχή. Υπάρχει επίσης η ανάγκη της απλοποίησης, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της διαδικασίες ε, πιστοποίησης. Ε, επίγουσα ανάγκη και αυτή. Τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και οι προθέσεις ε, μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά πρέπει ο Ευρωπαίος πολίτης να λάβει ισορροπημένες θέσεις που να σέβονται και τους μεγάλους παραγωγούς και τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι σήμερα ποινικοποιούνται και απαιτούν σαφείς και βέβαιες λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχετε το λόγο, κυρία Πασάτσου. Θα ακολουθήσει Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτού του σημαντικού κανονισμού. Θα έχουμε το χρόνο βέβαια να μπούμε στις λεπτομέρειες ε, κάθε θέσης, ε, αλλά σήμερα το πρωί θέλω να αναφερθώ ε, στον κανονισμό για την υγεία των ζώων και θέλω να τονίσω κάποιους γενικότερους στόχους που περιγράφησαν εδώ και που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εντάξει, καλά, καλή βέβαια η γενική στόχη, αλλά και οι λεπτομέρειες θα απαιτήσουν όλη την προσοχή μας για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτό που λέχθηκε για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου η οποία πρέπει να επιτευχθεί χωρίς ε, να μειωθεί βέβαια η ασφάλεια και η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Ε, πρέπει πραγματικά μεγάλη προσοχή να δώσουμε και κάθε δυνατή προσπάθεια να καταλάβουμε για να δώσουμε στους μεταποιητές, στους καλλιεργητές και όλους όσους δραστηριοποιούνται ε, στην αλυσίδα τις υποχρεώσεις τους και τις ευθύνες τους. Υπάρχει επίσης η ευθύνη των εθνικών, τοπικών και κοινοτικών αρχών. Ε, σημαντικό είναι να μπορούν όλοι να εργάζονται με την άνεσή τους, αλλά μέσα από την απλοποίηση της διαδικασίας δεν πρέπει να αφαιθούν απ' έξω ούτε δημόσιες αρχές. Ε, γιατί όταν θα κληθούν να, εφαρμόσουν την πολιτική για την υγεία των ζώων, ε, ε, δεν πρέπει να υπάρχει το, το άλοθη της περίπλοκης διαδικασίας. Ο άλλος σημαντικός στόχος που θέλω να τονίσω είναι η εξασφάλιση στους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές και όχι μόνο στους Ευρωπαίους ε, προϊόντα διατροφικά τα οποία καλύπτονται από εχέγγυα όσο αφορά την υγεία και την ποιότητα των προϊόντων. Αυτό είναι βασικό, θεμελιώδες. Ιδίως και σε σχέση με τον τρίτο στόχο που θέλω να τονίσω και ο οποίος είναι Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τρίτος στόχος που θέλω να αναφέρω να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που προέρχονται από τη ζωική παραγωγή ε, είναι πλήρως εμπορεύσιμα, όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως προς τρίτες χώρες, ε, προς του, οι ε, εμπορικοί μας εταίροι, πιο σημαντική. Πολύ σημαντική λοιπόν η εταίρεια αυτή για τα χαρακτηριστικά και ποιοτικά προϊόντα μας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στον τομέα της υγείας των ζώων για να ξεπεράσουμε και τα διασμολογικά εμπόδια που τίθενται από τους εταίρους μας. Μετά από 15 χρόνια οι Ηνωμένε Πολιτείε άνοιξαν την αγορά τους και σε κάποια αλλαντικά που παράγονται σε Ιταλικές περιοχές ε, ωστόσο, ε, σε, για συγκεκριμένους τομείς όπως η Σικελία, ε, για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που καλύπτουν το 30% της παραγωγής, παρουσιάζουν προβλήματα και δεν μπορούν να διατεθούν άνετα στις διεθνείς αγορές. Και υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι αυτοί οι στόχοι λοιπόν να εκπληρωθούν με πλήρη σεβασμό και στην πολιτική συνοχής, που είναι και καθημερινό θέμα συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο. Τέλος, η πρόταση κανονισμού παραπέμπει σε κάποιους χρόνους, ε, κάποιο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης σε σχέση και με τις ασθένειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το νομοθετικό αυτό πλαίσιο. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να εμβαθύνουμε και στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και μετά κύριος Γιάρ και τελευταίος θα είναι. Μαγκίνεση Είμαι πάρα πολύ σύντομη, επειδή είναι δύσκολο να κάνουμε τώρα μια αναλυτική συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους της Κομισιόν που έχουν εργαστεί πολύ σκληρά. Θα ήθελα και εγώ να πάω σε αυτή τη διάσκεψη τον Ιούνιο, αλλά από ό,τι μας είπαν ε, είναι στο Στρασβούργο η Ολομέλεια τότε και θα έχουμε και διάλογο για τις άμεσες πληρώμες, άρα δεν θα μπορέσουμε. Τώρα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο κάναμε μια συζήτηση χθε και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, βρεθούν πιο απλοί, εύκολοι τρόποι, ίσως ε, εκ των προτέρων επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο και να μην τα ακούμε εκ των υστέρων. Έχω ένα βασικό ερώτημα. Ο εξορθολογισμός, η συμπίκνωση, η μείωση του αριθμού των νομικών ε, μέσων μου αρέσει. Όμως, σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα τι διαφορά θα κάνουν αυτές οι προτάσεις σε αυτούς τους τέσσερις βασικούς τομείς. Αυτό ήθελα να μου Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, έχω να κάνω μια γενική φύσεως παρατήρηση που ισχύει για όλες τις εκθέσεις. Το έχουμε δει πολλές φορές. Η Κομισιόν προετοιμάζει οδηγίες και κανονισμούς και ξαφνικά ξεσπάει καβγάς στην κοινή γνώμη και εμείς ιδέα δεν έχουμε πάρει. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Ε, το είδαμε παλαιότερα στις ε, παραχωρήσεις, τώρα το βλέπουμε πάλι στους ε, σπόρους. Οι ασκούντες κριτικοί είναι καλύτερα ενημερωμένοι και τελικά ίσως θα μπορούσε κανείς να άρει πολλές επιφυλάξεις ε, γιατί αυτές οι επιφυλάξεις ε, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στους ε, κανονισμούς. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι εξή. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι, εντάξει, στην επικεφαλίδα αναφέρεται σπόροι και εμεί αυτό θέλουμε. Ε, θέλουμε οι απαρχιωμένοι κανονισμοί να συγχωνευτούν, να εναρμονιστούν, αλλά εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν μιλάει για εναρμόνιση και απλούστευση και προκύπτει το αντίθετο. Άρα και εδώ πρέπει να βρούμε ε, κάποια μορφή επικοινωνίας. Και εμεί θέλουμε με την εναρμόνιση να μην προκύπτει ε, γραφειοκρατία Όσον αφορά το δίκαιο περί σπόρων, τις νομοθετικές διατάξεις, ε, εγώ ήθελα να πω αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ που με εξέπλησε. Η συμμαχία που προκύπτει ανάμεσά μας είναι περίεργη, πρέπει να είμαστε και δυο προσεκτικοί. Λοιπόν, ε, πρέπει να έχουμε πράγματι την ελευθερία μετακίνησης των σπόρων, συμφωνώ και εγώ απόλυτα και απλά θέλω να επισημάνω στην Κομισιόν ότι και για το θέμα αυτό ε, θα κάνουμε προσεκτικούς ελέγχους. Ε, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με το μέγεθος της επιχείρησης για να μην καταλήξουν οι σπόροι σε λίγα μονοπόλια. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τη φύση, ούτε για τη γεωργία και σε τελική ανάλυση ούτε για την οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ε, Νομίζω ότι ακούσαμε τις παρεμβάσεις. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι άλλο από πλευρά της Επιτροπής. Αν δεν έχετε τίποτα άλλο το σημαντικό να πείτε, κλείνει αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξης, τελειώνει μάλλον. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι συμφωνήσαμε ότι πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων και ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους αδύναμους κρίκους ε, της αλυσίδας των τροφίμων. Να προστατεύσουμε τις περιφερειακές αγορές, τα περιφερειακά προϊόντα, Επίσης ε, πρέπει να προστατεύσουμε και τις ε, μικρότερες επιχειρήσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποικιλομορφία είναι ε, σημαντική για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και επανερχόμεθα στο σημείο υπαριθμών 13 που λέει «Ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής». Από την τελευταία συνεδρίαση έλαβαν χώρα τρεις διάλογοι, επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος, αλλά υπολείπονται ακόμα πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς ε, λοιπόν ε, συμμετείχαμε στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο ε, και είχαμε και μια άτυπη ανταλλαγή απόψε. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ως προς το ότι ο τριμερής διάλογος ε, που γίνεται σε τακτά διαστήματα ε, είχε το εξή χαρακτηριστικό. Όλοι θέλαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Συμφωνήσαμε στα λιγότερο σημαντικά ζητήματα, ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν πολιτικές ουσιώδεις αποκλήσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά στην Επιτροπή Γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω τη θέση του Συμβουλίου. Χθες ήταν σαφής η του Συμβουλίου. Με βάση αυτά που συζητήθηκαν ε, στο ε, Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, ε, δεν ε, θέλουν να τα ξανασυζητήσουν αυτά τα θέματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά τη οργανική συνεργασία και πρόκειται και για παραβίαση τη συνθήκη Λισαβόνα για εμά. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό πάρα πολύ σοβαρά στην Επιτροπή μα. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Ιρλανδό Υπουργό Γεωργία και θα μάλλον θα συναντηθούμε και θα του επιστήσουμε την ε, προσοχή στο πόσο σοβαρή είναι αυτή η κατάσταση. Βέβαια πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, όπως μέχρι τώρα. Θα σεβαστούμε ε, αυστηρά και μέχρι και την εντολή μας. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω αν έχουν ερωτήσεις ή να δισκεδάσω απορίες τους και αμφιβολίες τους ο Πρόεδρος. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή κύριο Μισελ Νταντά. Μας είπατε να είστε σύντομοι. Εγώ συμφωνώ ε, επιλέξει με ό,τι είπε ο Λουίς. Και είμαι και εγώ στη διάθεση των συναδέλφων για να απαντήσω σε ερωτήσεις τους. Μάλιστα, άρα ε, έκτακτα. Ε, μέχρι τώρα Εξαιρετικά τα ακούω. α ακούσω με τους υπόλοιπους. Κύριε Ράιμερ. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, να πω το εξής, ότι εμένα με φοβίζει ε, όλο και περισσότερο το ότι δεν θα τόσο με την ουσία αλλά με τις ισορροπίες ε, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Δηλαδή τελικά αγωνιζόμαστε αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας που όλοι επέγραψαν ε, πώς θα εφαρμοστεί. Εδώ όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι η γεωργία και επιτέλους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει ε, να αποφασίσουν να εφαρμόζουν στην πράξη τη συνθήκη της Λισαβόνας την οποία προσυπέγραψαν. Γι' αυτό προκύπτει αυτή η καθυστέρηση στις ε, διαπραγματεύσεις. Θα ήταν λοιπόν πολύ συμπαθητικό, όπως σας είπα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιτέλους να εφαρμόζουν τη συνθήκη της Λισαβόνας στην πράξη. Πρόεδρος, ε, ε, πράγματι, σωστά τα είπατε, συμφωνούμε απόλυτα. Ο κύριος Χόισλινγκ. Κοιτάξτε, ε, βέβαια οι φιλελεύθεροι είναι μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού. Ε, μήπως θα πρέπει λοιπόν ε, να τοποθετηθούν εδώ τα κόμματα γιατί δεν είναι δυνατόν ως ε, κοινοβούλιο όπως ε, ελέγχεται χθες ε, στον τριμερή διάλογο να λέμε ότι αυτό το έχουν διαπραγματευτεί αρχή κρατών και κυβερνήσεων και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση όταν πρόκειται ας πούμε για τον καθορισμό ανώτατων ορίων ή για το, για το δεύτερο πυλώνα αυτό είναι προσβολή του κοινοβουλίου διότι όταν οι αρχηγοί κρατών καταλήγουν καταλήγουν ε, σε θέματα γεωργικής πολιτικής. Πρόκειται κατ' ουσίαν για συμβιβασμούς. Σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών είπε ότι πρέπει να βρούμε κάποια απάντηση. Βεβαίως και πρόκειται για ε, διαφωνία ανάμεσα σε θεσμούς. Η κυρία Μέρκελ λέει δεν θέλουμε περικοπές και ξαφνικά ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κατ' ουσίαν εντολή προς το Κοινοβούλιο. Εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει οι φιλελεύθεροι θα ε, μιλήσουν στο Κοινοβούλιο και θα πούνε στην κυρία Μέρκελ ότι οι αρμοδιότητες ε, για τη γεωρική πολιτική αφορούν και και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα αυτήν την Επιτροπή. Πρόεδρος, κοιτάξτε, στις Βρυξέλλες είμαστε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι λίγο σουρεαλιστικό να πρέπει να καλύψουμε τέσσερα θέματα το ένα μετά το άλλο, να θέσουμε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή να μην έχει το δικαίωμα να μας απαντήσει. Τώρα, η έκθεση για τον τριμερή διάλογο. Έχω μια πρόταση. Είμαι υπεύθυνο για μια έκθεση για την εξυγχρονισμό των ε, δημόσιων συμβάσεων για την εσωτερική αγορά ε, ε, ε, τώρα ο τρόπος που λειτουργούμε είναι να ζητάμε μια εντολή και μετά να την χρησιμοποιούμε για να διαπραγματευτούμε. Ε, ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εξ αρχής να είμαστε ρεαλιστές ως προς το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ε, δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε όλη την ώρα τριμερή διάλογο και μετά να χανόμαστε στις λεπτομέρειες γιατί πρόκειται για πολιτικές πάρα πολύ περίπλοκες. Ε, προτείνω, δεν έχω ίσως την εξουσία να το κάνω, αλλά μπορώ να το πω, να ξεκινήσουμε συστηματικά στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Γεωργίας να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για το πού είναι ο τριμερής διάλογος εκτός μικροφώνου το υπόλοιπο της παρέμβασης. Ε, ίσως ε, μπορείτε να επαναλάβατε αυτό που είπατε στο τέλος, γιατί είχε κλείσει το μικροφωνό σας. Έλεγα ότι ίσως η πρότασή μου έρχεται πολύ αργά γιατί θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο αλλά είπε ότι ίσως θα μπορούσαμε ε, σε περίπτωση παράτασης, αλλά και γενικά σαν Επιτροπή Γεωργίας το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, είτε απόγευμα είτε πρωί, να είναι ο απολογισμός για τον τριμερή διάλογο και να παρουσιάζουν οι εισηγητές στην αρχή της κάθε συνεδρίασής μας τι έχει γίνει. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δώσαμε το λόγο σε όλους όσοι τον ζήτησαν. Ε, θα ξανασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα, να πω κάτι για τις επόμενες συνεδριάσεις που θα γίνουν στις 29 Μαΐου. Ε, 19 Ιουνίου και 20 Ιουνίου, με συγχωρείτε. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και θα τα ξαναπούμε στι 19 ε, Ιουνίου από 3 μέχρι 6.30 και 20 Ιουνίου από 9 μέχρι 12.30. Γεια σα. bye